Cari colleghi, diamo inizio alla... Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε το τμήμα της ε, συνεδρίας μας που αφορά τις ψηφοφορίες. Πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, μπορώ να σας ανακοινώσω ότι η Οικονομική Επιτροπή διαβίβασε μια τροποποίηση στο κείμενο που διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα δημοσιευθεί η τροποποίηση, η διόρθωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 4 του εσωτερικού κανονισμού, η διόρθωση αυτή θεωρείται εγκεκριμένη εκτός εάν εντός 48 όρου μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 βουλευτές δεν επιθυμούν να τεθεί σε ψηφοφορία.